So, dear colleagues, I think we should start. νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα έπρεπε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και θα τα πω από εδώ και πέρα στα γερμανικά. Να μην τιμωρήσουμε αυτούς ε, που είναι στην ώρα τους, οπότε ξεκινώ. Και όπως πάντα ξεκινούμε με το σημείο της ημερήσια διάταξης που είναι η έγκριση του σχεδίου ημερήσια διάταξης. Μόλις ε, μάθαμε ότι η συζήτηση με τους δύο επιτρόπους Ναύρατσιτς και Έτιγκερ πρέπει να αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη. Διότι δεν ε, υπάρχει χρόνος για σήμερα, όπως μας είπαν, αλλά υποσχέθηκαν κάποια στιγμή σύντομα να βρούμε μια νέα ημερομηνία. Θα περιμένουμε να δούμε. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε δεκτό το σχέδιο της Μερσίας Διάταξης όπως τροποποιήθηκε ή έχετε εσείς να προτείνετε κάποια προσθήκη αλλαγή. Όχι, επομένως εγκρίνεται όσο έχει η ημερήσια επομενως εγκρινεται οσο εχει η μερσια διαταξη και περνάμε στο σημείο 2 έγκριση των πρακτικών. Έχετε το σχέδιο πρακτικών της συνεδρίας επιτροπής μας στις 22 Οκτωβρίου. Παρατηρήσεις. Δεν βλέπω, οπότε ως ήθιστε προτείνω να θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά εγκρίνονται αν δεν υπάρξει κάποια παρατήρηση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αυτής. Έτσι θα προχωρήσουμε λοιπόν. Ανακοινώσεις Προέδρου, τρίτο σημείο. Διερμηνία σήμερα έχουμε στα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα αγγλικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τσεχικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά, ρουμανικά. Και όπως πάντα σας επενθυμίζω πως η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών, 20 Νοεμβρίου, ε, τις λάβατε με email στις 22 Νοεμβρίου και θεωρούνται ότι εγκρίθηκαν γιατί μέχρι την ε, προθεσμία που είχαμε βάλει, 26 Νοεμβρίου δηλαδή, δεν λάβαμε καμία αντίρρηση. Επίση ε, να καλωσορίσω τον ε, Μπόγκουσλαφ Ζόνικα ως νέο μέλος Επιτροπής μας αντικαθιστά τον Μπόγκταν Βέντα που όλοι γνωρίζετε τυχερός ο ίδιος βέβαια έγινε δήμαρχος και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σίγουρα με δυσαρεστή που τον χάνουμε από συνάδελφο, αλλά δεν είναι εδώ ο μπόκους Μπόκου Λαυσόν για να τον καλωσορίσουμε, αλλά τέλο πάντων τον καλωσορίζουμε νοερός. Θα το τα πούμε την άλλη φορά. Και περνάμε στο σημείο 4 τη ημερήσιας διάταξη. Ε, έχουμε την ε, ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότηση για τη θέση του προγράμματο δικαιώματα και αξίες που βέβαια εμείς ε, έχουμε αγωνιστεί ως Πολιτισμού να έχουμε ε, δικαιώματα. Ε, και έχουμε εδώ το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Η συγγήτρια ήταν η Σιλβίγκη Γιόμ. Δεν ήταν και τόσο ομαλέ διαπραγματεύσει με τη λίγο θα θέλαμε από ό,τι ξέρω. Αλλά ε, στη συνέχεια των διαβλέψεων ελπίζω να βελτιωθεί κάπω η κατάσταση. Σιλβί, θέλει να πει κάτι. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ γρήγορα για να μην ε, επιμηκύνω και τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία στην Επιτροπή Πολιτισμού. Να ευχαριστήσω και την Γραμματεία για την υποστήριξη. Πολύ σωστά είπε. Ήταν πολύ για να τι χαρακτηρίσω έτσι, τη συζητήση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και το βασικό πρόβλημα, ελπίζουμε να μπορέσουμε να το λύσουμε, είναι ότι η Επιτροπή προσπαθεί να μειώσει ε, τη θέση του προγράμματος Ευρώπη των Πολιτών ε, στο νέο πρόγραμμα και γι' αυτό πρέπει να επαγρυπνούμε. Και ότι μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές ό,τι αυτή τη λειτουργία του προγράμματος, οι αδελφοποιήσεις ε, και η συμμετοχή των πολιτών μεταξύ άλλων, είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε και τους επόμενους ε, μήνες εν ώψη και των ευρωεκλογών. Θέλουμε να συνεχιστούν να ισχύουν και να μην μπουν σε κίνδυνο. Υπάρχει κάποια καλύτερη συνεννόηση τώρα με τη Λίμπε και ελπίζω ότι έτσι θα προχωρήσουμε μεταλλευόμενοι αυτό το θετικό, αυτή τη θετική εξέλιξη. Ευχαριστώ. Η ε, πρόεδρος, ευχαριστώ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Λίμπε και προσπάθησα να ξεκαθαρίσω ε, τη μεγάλη σημασία που έχει για μας ως Επιτροπή αυτό το πρόγραμμα, ελπίζοντας ε, να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει κάπως και τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε ευθύς αμέσως στην ψηφοφορία και ξεκινάμε με τη συμβαστική 1. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Ψήφι υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ψήφι πέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 και 155 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Πηγαίνουμε στην συμβιβαστική 8 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 απορρίπτεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά να το ελέγξουμε καλύτερα. 168. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 9 προς 7. 169 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 170 και 171 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω απορρίφθηκε να ελέγξουμε. 172. Πέρασα. Πράγματι, 10 κατά 6 υπέρ. Ε, συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 199. Υπέρ, κατά, αποχές, Ας ελέγξουμε την 199, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. ήταν 16 όλα. Μάλλον 16 όλοι είχατε ψηφίσει υπέρ. Αλλά δεν σηκώνετε τα χέρια, δεν έβλεπα. 200 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Τη 200. Geschlossen. Πέρασε. 9 ήταν η κατά, 7 υπέρ, άρα απορρίφθηκε. Η 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τέλο πάντων, να μάλλον ξανά, ποιοι είναι υπέρ της 203. Ποιοι είναι κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 217 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 220 υπέρ, 220 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 221 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 222 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 224 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε 224 Πέρας. Εννέα προς 8. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία της 44. Πέρας. 12 προς 4. Εγκρίνεται. Δεν το είχα καταλάβει. 45 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προπολογία 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 61. Geschlossen. Πέρας. 11 προς 6. Και αυτό δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων. Πάμε στην 21 συμβαστική υπέρ. Κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 70, άρχεται του ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρασε. 11 προς 6. Εγκρίθηκε. 22 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 84 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε την 87. Πέρασε. Απορρίφθηκε 9 προς 8. συμβιβαστική, 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίθηκε. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 25 συμβιβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 26 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται δεν κατάλαβα τι σημαίνει πράγματι αυτό το 8 από πάνω 113 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία που είναι ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 16 υπέρ μία αποχή. Ομόφωνα δεκτή λοιπόν. Συγχαρητήρια Σίλβια. Στη Σιλβή μάλλον. Και καλή επιτυχία στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων των δευλεύσεων με τη Λίμπε. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνεις ό,τι καλύτερο για μας. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξη. Πρόκειται για τον έλεγχο και την εξέταση των ψηφοφοριών που αφορά το πρόγραμμα εράσμος. Ο Μιλανσφέρη είναι εισηγητής. Έχουμε 684 τροπολογίες. Σήμερα ουσιαστικά θα κάνουμε κάτι που αν θέλετε είναι ένα μεταβατικό βήμα, για κάποιους αυτό είναι συνηθισμένο, γιατί υπάρχει μια πάγια συνήθεια σε άλλες επιτροπές, σε μας όχι. Ε, δεν εξετάζουμε αυτόν τον τρόπο τις τροπολογίες, συνήθως εδώ. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σας πω πριν ξεκινήσουμε ότι στις 22 Ιανουαρίου προβλέπεται η ψηφοφορία, η οποία όμως για να είναι επιτυχής θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως διαβούλευση και συμβιβασμός ε, για πολλά σημεία που αφορούν τροπολογίες. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε, αν θέλετε, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία στις 22 Ιανουαρίου και θα αναγκαστούμε να ψηφίσουμε στην αρχική ημερομηνία που ήταν το Φεβρουάριο, 22 Φεβρουαρίου. Θα δώσω όμως το λόγο στον εισηγητή, τον ε, Μίλαν Σφέρ, για να μας παρουσιάσει τις θέσεις του για τη τροπολογία. Σας ευχαριστώ. για τα πρώτα σας σχόλια, αγαπητοί σκιώδεις εισηγητές και μέλη της Επιτροπής. Όπως ανέφερε και, ο, και η πολλές από τις τροπολογίες έχουν υποβληθεί για το πρόγραμμα αυτό Erasmus Plus. 684 είναι ο συνολικός αριθμός αυτών των τροπολογιών την προηγούμενη Παρασκευή ήδη επεξεργαστήκαμε κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες και έχουμε προβλέψει επιπλέον συναντήσεις ε, με τους ε, σκιώδεις εισηγητές ε, για να μπορέσουμε και από κοινού με τους συντονιστές να προχωρήσουμε σε περαιτέρω συμβιβαστικές τροπολογίες για θέματα που αφορούν τους νέους, την κατάρτιση, τον αθλητισμό θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με τους κοιόδης συζητητές στο Στρασβούργο. Θα ακολουθήσει συζήτηση περαιτέρω θεμάτων και τομέων και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε την εργασία μας μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε όντως στις 22 Ιανουαρίου όπως έχει προβλεφθεί. Έχουμε προετοιμάσει συμβιβασμούς γύρω από κάποια θέματα τα οποία σας προανέφερα. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στη μέθοδο εργασίας μας και οι μέχρι τώρα συμβιβαστικές τροπολογίες ουσιαστικά προέρχονται από πολλές κοινοβουλευτικέ ε, ομάδες και ουσιαστικά οι περισσότερες πολιτικές ομάδες συμφωνούν με τον τίτλο Erasmus Plus και όσον αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό. Επίσης για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις, συμφωνούν οι περισσότερες ομάδες. Όσον αφορά την εσωτερική κατανομή των κονδυλίων, πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να βρεθεί συμφωνία και εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι θα πρέπει να υποβληθούν ε, τροπολογίες οι οποίες πλησιάζουν ε, με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άλλες ε, προτάσεις υπάρχουν που αφορούν άλλη κατανομή των κονδυλίων. Οι σοσιαλιστές προτείνουν μείωση των κονδυλίων για κάποιους τομείς, όπως παραδείγματο χάρη η δράση ζωμονέ και ο αθλητισμός. Πρόκειται για κονδύλια και δραστηριότητες που ουσιαστικά αυξάνουν την ε, συμμετοχή των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Το πρόγραμμα Ζώμων είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι τελικά οι απόψεις των ΜΕΝ και των ΔΕ δεν είναι εντελώς διαφορετικές και ότι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι περισσότερες ομάδες είναι σωστά προτείνεται ενδυνάμωση και ενίσχυση των σχεδίων και των προγραμμάτων τα οποία ευρείας βάσης και μικρά προγράμματα, μικρές εταιρικές σχέσεις, στήριξη μικρών ομάδων. Είναι κάτι που το προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης υπάρχουν κάποιοι ευρωβουλευτές, οι οποίοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστούν κάποιοι τομείς από το πρόγραμμα Εράσμους εάν δεν υπάρξουν αυτές οι συνεργασίες. Εγώ διαφωνώ. Πιστεύω ότι βεβαίως πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις συνεργασίες, όχι μόνο γιατί ε, προέρχονται από τη βάση, αλλά γιατί πραγματικά είναι αποτελεσματικές. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το θέμα της προστιθέμενης αξίας αυτών των προγραμμάτων. Ε, στηρίζουμε τις τοπικές αυτές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ αυτών των ε, τοπικών δραστηριοτήτων. Δεν μπορούν όλες οι δραστηριότητες να είναι υπερεθνικές και να συμπεριλαμβάνουν περισσότερες χώρες. Θα πρέπει και κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες που θα στηρίξουμε να έχουν τοπική βάση. Και πιστεύω ότι το πρόγραμμα Erasmus Plus βεβαίως πρέπει να δείξει ότι ε, υπάρχει σε όλες του τις πτυχές προστιθέμενη αξία, αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και κάποιες διαφορετικές διατυπώσεις έτσι ώστε να βρεθεί συμβιβαστική λύση στα σημεία αυτά που ακόμα εκκρεμούν. Πιστεύω επίσης ότι το θέμα της εικονικής κινητικότητας και της εικονικής δραστηριότητας θα πρέπει να διευκρινιστούν. Δηλαδή, μεταξύ της πραγματικής κινητικότητας και της εικονικής δραστηριότητας θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής διάκριση. Παρ' όλα αυτά, στηρίζουμε τις εικονικές δραστηριότητες, αλλά θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη σαφήνεια στον ορισμό αυτών των εικονικών, δραστηριοτήτων. Επίσης, η εκμάθηση γλωσσών με την βοήθεια νέων τεχνολογιών και η εκμάθηση γλωσσών επιτόπου στην ε, χώρα που ομιλείται η γλώσσα αυτή. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να μάθει κάποιος μία ξένη γλώσσα. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τις ειδικέ ανάγκες των συμμετεχόντων. Όσον αφορά την καταπολέμηση του αποκλεισμού. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και έχω συμπεριλάβει κάποια άρθρα που αναφέρονται ακριβώς σε αυτό το θέμα, την καταπολέμηση των αποκλεισμών, του αποκλεισμού. Υπάρχουν και οι ορισμοί των ατόμων με λιγότερες δυνατότητες και ευκαιρίες. Τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης και τι αντιμετωπίζεται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τη συμμετοχή κάποιων ατόμων στο πρόγραμμα Erasmus+. Εδώ ένα καθοριστικό σημείο είναι το θέμα της ε, χρηματοδότησης της κινητικότητας και το βιωτικό επίπεδο στην κάθε χώρα. Το θέμα των αμοιβών, των αποδοχών για την ε, εργασία. Ίση εργασία, ίσες αποδοχές. Αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά αντιτίθεται στον κύριο στόχο αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή η χρηματοδότηση, αν θέλετε, της κινητικότητας στα επίπεδα της κάθε χώρας σίγουρα θα βοηθήσουν να εξοδοτερεθούν οι διαφορές στο επίπεδο που δυστυχώς υπάρχει από τη μια χώρα στην άλλη. Καταλαβαίνετε ότι αν δοθεί η ίδια χρηματοδότηση για κάποιον που σπουδάζει στη Φιλανδία και για κάποιον που σπουδάζει στη Ρουμανία, αυτό δεν είναι δίκαιο. Και ουσιαστικά θα αποθαρρύνουμε κάποιους οι οποίοι θα θέλανε να συμμετάσχουν στο Erasmus Plus. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί λοιπόν ο στόχος μας να είναι κάτι τέτοιο. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα στηρίξω καμία τροπολογία που πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορώ να στηρίξω απολύτως καμία τροπολογία που να ζητάει τέτοιου είδους συμμετοχή που θα δίνει δηλαδή πλεονέκτημα σε αυτούς που είναι στη Νότια ή στη Βόρεια Ευρώπη. Όσον αφορά την κινητικότητα λοιπόν, Ο πολλαπλασιασμός των κονδυλίων που εκατονταπλασιάζονται όσον αφορά παραδείγματος χάρη την κατάρτιση των ε, καθηγητών, ιδιαίτερα για τον ε, τομέα του αθλητισμού. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι αθλητές, οι επαγγελματίες αθλητές πολλές φορές έχουν πάρα πολύ βραχυπρόθεσμες σταδιοδρομίες και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όσο περισσότερους μπορούμε μέσω αυτών των προγραμμάτων κατάρτισης στην κατηγορία 1. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε και ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες και πολύ ελλειπή προσόντα. Γι' αυτό και σας προτείνω να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι κατηγορίες ε, στην ε, δράση κλειδί υπαριθμών 1. Όπως βλέπετε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλες χώρες αυτό το πρόγραμμα, τρίτες χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιες εθνικές και πιο ολοκληρωμένες προκλήσεις. Κυρία Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον Μάρκο και την Πέτρα που με στήριξαν στην προετοιμασία αυτή τη έκθεσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης για όλη σας την προσπάθεια για τις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μίλαν. Εδώ κανονικά θα έδινα το λόγο στην Κριστίνα Λιμπάτσκα. Βλέπω όμως ότι έχει αφιερώσει όλη της την προσοχή στην οικογένειά της αυτή την εποχή. Γι' αυτό και θα δώσω το λόγο στην Σίλβια Κώστα, η οποία πιστεύω ότι σαν ε, συντονίστρια θα πάρει το λόγο. Στέλνουμε όλες μας τις σκέψεις και τις ευχές στην Κριστίνα, η οποία περνάει μια πολύ δύσκολη στιγμή και ελπίζω πολύ γρήγορα να επανέλθει εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ όλους για την συνεισφορά τους, όλους τους βοηθούς, τη γραμματεία. Έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά με τα πρώτα αυτά συμβιβαστικά, τις πρώτες αυτές συμβαστικές τροπολογίες, τις οποίες συμφωνήσαμε. Δεν θέλω τώρα να μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Το κάναμε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά πρέπει να σας πω ότι και εγώ παρακολουθώ το θέμα πολύ στενά. Το θέμα τώρα της κατανομής, της χρηματοδότησης, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν βασικές διαφορές και ότι υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί μία κοινή αν θέλετε, στάση με κάποια ποσοστά πάνω, κάποια κάτω, αλλά νομίζω ότι οι προτάσει όλων είναι μάλλον λογικές ε, για τα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα Ζωμονέ όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση. Μέχρι τώρα τα μέτρα στο πρόγραμμα Ζωμονέ ήταν ξεχωριστά και στόχευαν ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να συμπεριλάβουμε τα μέτρα ζωμονέ στην γενικότερη επαγγελματική κατάρτιση. Το νέο άρθρο 7 ουσιαστικά, έτσι όπως έχει διατυπωθεί, συμπεριλαμβάνει αυτές τις σπουδέ που αφορούν τα ευρωπαϊκά θέματα και έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για πολύ συγκεκριμένες σπουδέ που αφορούν την Ευρώπη. Εδώ δεν ξέρω μου φαίνεται λογικό να υπάρχει ξεχωριστή χρηματοδότηση και άλλος ε, προϋπολογισμός. Τώρα, για τις ε, επιχορηγήσεις 3,4% για τις εθνικές υπηρεσίες. Αν παραμείνουμε εκεί που είμαστε και να μην μειωθεί εδώ αυτό το ποσοστό σε 3,2%, αυτό προτείνει η Επιτροπή. Έχω την εντύπωση ότι με δυσκολία θα εξηγήσουμε στις ε, εθνικούς οργανισμός ότι πρέπει να αναλάβουν περισσότερες δραστηριότητες, περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά λιγότερη χρηματοδότηση. Εγώ προτείνω να παραμείνουμε στο 3,4%. Έχουμε και μια ολόκληρη σειρά νέων προγραμμάτων ε, που συμπεριλαμβάνονται στο Erasmus+. Plus. Πρόκειται για σχέδια τα οποία ουσιαστικά τα περιγράφουμε σαν ε, μαύρα κουτιά 40 δις ουσιαστικά ε, έχουμε κατά κάποιο τρόπο προβλέψει. Αμφιβάλλω αν θα υπάρξουν αυτά τα ποσά. Θα δούμε τελικά ε, αν τα ποσά αυτά συγκεντρωθούν. Αν όχι, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αμφισβητήσουμε κάποια από αυτά τα νέα σχέδια. Και εδώ βεβαίως, ε, αν θέλετε, συμπεριλαμβάνονται διάφορα προγράμματα κατάρτισης επαγγελματικής, θέματα ακαδημαϊκών προγραμμάτων, πανεπιστημιακών, αριστείας. Έχω την εντύπωση ότι κάποια από αυτά τα ε, σχέδια και προγράμματα περιγράφονται με ένα κάπως ε, σαφή τρόπο τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια παραδείγματο χάρη. Προς το παρόν υπάρχει μια πειραματική, πιλωτική φάση, αν θέλετε, όσον αφορά αυτά τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ας περιμένουμε να ολοκληρωθεί για να δούμε όταν υπάρξει η ολοκλήρωση αυτής της πιλωτικής φάσης και η αξιολόγησή της, να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ακριβώς θα προκύψει. Εγώ πραγματικά έχω συζητήσει με ειδικού, με καθηγητές, με ακαδημαϊκούς και δεν έχω καταλάβει με σαφή τρόπο τι ακριβώς είναι αυτή η έννοια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημιακό Ανώτατο Ίδρυμα Ευρωπαϊκό, γιατί έχω ακούσει πολύ διαφορετικές απόψεις. Discover EU, ανακάλυψε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία η οποία πρέπει να στηριχθεί, είναι εξαιρετικά σημαντική να ανακαλύψει κανείς τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ αυτή η πρωτοβουλία κατά την άποψή μου θα πρέπει να διασφαλιστεί με νομοθετικό κείμενο, είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται με το ευρωπαϊκό πολιτιστικό έτος, με τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα κτλ. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν. Θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κινδυνεύσουμε να χάσουμε αυτήν την ε, πρωτοβουλία, ιδιαίτερα εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την ε, χρήση των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων, των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογούμενων. Α, εδώ νομίζω όμως ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απλουστευτούν. Συνεχίζει να είναι δύσκολη η πρόσβαση σε κάποια προγράμματα, γι' αυτό και μιλάμε για απλές διαδικασίες, για απλουστεύσεις διαδικασιών, για αλληλεγγύη, για καταπολέμηση του αποκλεισμού, για συνοχή. Το πρόγραμμα Εράσμους, λοιπόν, μπορεί να συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις προτάσεις ίση αμοιβή, ίσες αποδοχές για, ίση, για ίδια εργασία. Εδώ θα πρέπει σαφώς να κοιτάξουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προετοιμάσει την πρωτοβουλία αυτή. Θα πρέπει να ενημερωθούν οι συνεργάτες έτσι ώστε όντως να βρεθεί μια λύση που να ανταποκρίνεται στο πραγματικό βιωτικό επίπεδο της κάθε χώρας. Το θέμα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Και εδώ θα πρέπει λίγο να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτή την ιδέα. Σε όλα τα προγράμματα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, κάθε φορά προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να την ενισχύσουμε με μία, αν θέλετε, προσεκτική κωδικοποίηση των ε, προγραμμάτων, έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάνω από 20 διαφορετικοί ορισμοί του τι είναι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια και όχι περισσότερη ασάφεια αν θέλετε. Πρέπει να βρεθεί μια καλή ε, λύση όσον αφορά το ποιος είναι αυτός ο ορισμός της ε, προστιθέμενης ευρωπαϊκής αξίας. Και πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να προετοιμαστούμε για μία μάχη με το Συμβούλιο όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων και αν δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Τι θα μπει και τι θα βγει, τι θα μείνει απ' έξω από το Erasmus Plus. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε όλους τους σκιώδεις, αλλά δεν είναι όλοι εδώ. Ο Τζιλ Εύανς έχει το λόγο. Α, ή ε, κυρία Εύαν, συγγνώμη. Thank you very much, Chair, and can I thank the uh, rapporteur. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή γιατί ιδιαίτερα συμπεριέλαβε μερικές από τις δικές μου τροπολογίες τις συμβαστικές ως προς την ε, αύξηση της ε, απομάκρυνσης, μάλλον την απομάκρυνση από τους αποκλεισμούς και τη γενικότερη ενσωμάτωση. Ξέρετε ότι ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι οι νέοι θεωρούν ότι όλο αυτό το πλαίσιο δεν είναι προσπελάσιμο για τους ίδιους. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, δούμε και τις οργανώσεις υποστήριξης και ένα ευρύτερο φάσμα συμμετοχών στο Εράσμους και ιδιαίτερα συμμετοχή ανθρώπων με αναπηρίες ΛΟΑΔ ή αυτών που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες. Αυτό αφορά και το Erasmus Plus. Υπάρχουν ανησυχίες ως προς τη χρηματοδότηση του κόστους των ανταλλαγών. Γι' αυτό υπέβαλα τροπολογία έτσι ώστε να υπάρχει χρηματοδοτική υποστήριξη. Η Ρέτζη μίλησε για το κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής και αυτό θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Επίσης έχει μεγάλη σημασία η εκμάθηση γλωσσών που είναι αναπόσπαστο τμήμα του Εράσμους. Αλλά αυτό αφορά, θα πρέπει να αφορά και την νοηματική και τις γλώσσες των μειονοτήτων έτσι ώστε να προωθήσουμε και την δίγλωση και πολύγλωση εκπαίδευση και τα έγγραφα να είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες των συμμετεχόντων καθώς και γλώσσες που δεν είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο θέμα που αφορά την γλωσσική ισότητα αφορά την χρήση των ε, τεχνολογιών ε, εχμής, έτσι ώστε να ε, χρησιμοποιήσουμε και τις συνέργειες με τον ορίζοντα της Ευρώπης και να υπάρχει και αυτόματη μετάφραση μέσα στα πλαίσια του προγράμματος. Αυτό καλύπτεται και από την πρώτη συμβιβασμού. Επίσης υπέβαλα τροπολογίες έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι πιο ανοιχτό. Ο εισηγητής θέλει να το κάνει στο μέτρο του δυνατού. Εγώ ε, εκπροσωπώ την Ουαλία που συμμετέχει ενεργά στο Erasmus Συν και υποδεχόμαστε πολλούς φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε και στο μέλλον ε, τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, ό,τι και να συμβεί μετά του, το Μάρτιο του επόμενου έτους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για εμάς, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί μας επισκέπτονται πολύ συχνά. Ως προς τον προϋπολογισμό έχω υποβάλει μία τροπολογία, γιατί για το πρώτο έτος θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το κόστος είναι υψηλότερο σε σχέση με το τελευταίο έτος του 2020. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και η επαγγελματική κατάρτιση ως προς τη, ε, το θέμα της βάσης, της υποστήριξης από τη βάση. Αυτό το έθιξα και σε ορισμένες τροπολογίες μου. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε προγράμματα ευρείας κλίμακας. Μιλώ για τοπικά προγράμματα και ε, προγράμματα υποστήριξης ε, σε σχέση με την υγεία και τη διαβίωση και ούτω καθεξής. Θα το δούμε αυτά στη συμβιβαστικές στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο, αν θέλει βέβαια. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κύριε Τσβέρ για την εργασία σας. Για τον κανονισμό του Ερασμού. υπάρχουν πολλές τροπολογίες και εκτιμούμε την, την όλη εργασία για να φτάσουμε σε μία συμφωνία. Επίσης, το ε, πρόγραμμα του Κοινοβουλίου είναι φιλόδοξο και όλες οι τροπολογίες που έχουν ε, υποβληθεί αφορούν ε, την κοινή διάρθρωση του προγράμματος. Πρόκειται για ένα εικονικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα θέλαμε να είναι πιο ανοιχτό και πρόγραμμα που να τίνει προς την ενσωμάτωση, γι' αυτό θα θέλαμε να τίνουμε σε αυτό τον στόχο ως προς τις προθέσεις μας και τις ε, τροπολογίες που έχουν ε, υποβληθεί, πώς συσχετίζονται ως προς την απλούστευση. Αυτό είναι ένα βασικό μας ε, μέλημα έτσι ώστε να υπάρχει μία οριζόντια ίση προσέγγιση και μιλάμε για εκδήλωση ενδιαφέροντος από όλους μέσα στα πλαίσια του εγχειρήματος διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους. Θεωρούμε ότι ορισμένες τροπολογίες ίσως αντιβαίνουν σε αυτή την τάση απλούστευσης. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ε, στοχοθέτησης και βασική χρηματοδότηση. Θα μπορούσε να υπάρχει επιπρόσθετο άχθος του συμμετέχοντες και νομίζω ότι το πρόγραμμα ε, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες ανάγκες της επταετίας. Το θέμα της ενσωμάτωσης το θίξατε και εσείς. Μιλάμε για συγκεκριμένες ομάδες, ε, στόχους ή οργανώσεις και θα θέλαμε να υπάρχει υψηλός βαθμός ενσωμάτωσης. να έχουμε καλύτερη ε, διοργάνωση και οργάνωση των δράσεων, καλύτερη συμμετοχή της βάσης και κινητικότητα, καθώς και μεθόδους ευέλικτης ε, κινητικότητας για να μην υπάρχει επιπρόσθετο διοικητικό άχθος. Επίσης, τα μέσα αυτά θα πρέπει να είναι φιλικά προς το χρήστη και θα θέλαμε οι οργανώσεις βάσης να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε όλα τα σχέδια Εράσμους και να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση ως προς τους ε, δικαιούχους και τις εθνικές οργανώσεις. Επίσης, στις τροπολογίες τονίσατε ότι το ετήσιο πρόγραμμα είναι ε, μία κατευθυντήρια γραμμή και αυτό αφορά και τις ε, κατεξιδότηση πράξης ως προς τις δράσεις εκπαίδευσης αυτό όμως αντιβαίνει το άρθρο 291 της συνθήκης. Ξέρετε ότι τα ετήσια προγράμματα θα πρέπει να συμβαδίζουν με το ακαδημαϊκό έτος, έτσι ώστε οι φοιτητές και οι καθηγητές να μπορέσουν να προγραμματίσουν την κινητικότητα αυτή και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους νέους σε αυτή την κινητικότητα. Έχει σημασία λοιπόν ο χρονισμός, γιατί η κατεξιοδότηση ε, πράξης είναι χρονοβόρες. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό θα ήταν επιζήμιο προς τις ομάδες στοχοθέτησης ως προς το, την ονοματοδοσία του προγράμματος θεωρούμε ότι είναι αρκετά γνωστό. Είχαμε και την πανηγυρική επέτειο και νομίζω ότι όλοι κατανοούν ότι το Εράσμους καλύπτει όλους τους τομείς και όχι μόνο την ανώτατη εκπαίδευση. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αλλάξει η ονομασία. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα ζητήματα. Μιλήσατε για ίση αμοιβή, για ίση εργασία, για τους ερευνητές, καθηγητές, διδακτικό προσωπικό και ούτω καθεξής. Αλλά εδώ Μιλάμε για επιστροφή δαπανών και όχι μισθούς καθεαυτούς. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και να δούμε τεχνική υφής ζητήματα και τις επόμενες ημέρες θα ξαναδούμε τις τροπολογίες και τις συμβιβαστικές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και θα ε, συνεχίσουμε να σας ε, βοηθάμε σε αυτό σας το εγχείρημα έτσι ώστε οι δικαιούχοι να έχουν ακόμα περισσότερα πλειονεκτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την απλοποίηση των προγραμμάτων, νομίζω ότι χρειάζεται και η Επιτροπή να κάνει κάποιες προσπάθειες Έχουμε το θέμα του παραδείγματος των εθνικών οργανισμών και υπηρεσιών. Όλα τα προγράμματα, ο τρόπος που πρέπει να παρουσιαστούν και να υποβληθούν. Έχει τριπλασιαστεί το κείμενο αυτό που πρέπει να υποβληθεί. Ήταν δύο σελίδες και τώρα είναι έξι σελίδες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι απλοποίηση. Αυτό είναι κάνουμε τα θέματα πιο περίπλοκα από ό,τι ήταν. Και δεν είναι ο σκοπός μας αυτός. Και θα ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν ήσασταν ε, παρούσα στη συζήτηση που είχαμε για την, ε, τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης. Δεν έχουμε κανένα θέμα να περνάμε από αυτήν την μέθοδο από τη στιγμή που πρόκειται για την τεχνική εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων, τεχνική υλοποίηση αν θέλετε. Καθαρά όμως αυτό, όταν πρόκειται όμως για πολιτικές προτεραιότητες που πρέπει να θεσπιστούν, όταν πρόκειται για προγράμματα εργασιών τα οποία πρέπει να οργανωθούν και να γίνουν από εμάς την νομοθετική αρχή, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουμε την συμμετοχή μας μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να περάσει σαν μήνυμα και στους επικεφαλείς ε, των ε, διευθύνσεων και στους επιτρόπους. Εάν θέλει η Επιτροπή περισσότερη ευελιξία, είμαστε σύμφωνοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι τομείς αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να διεκπαιρεωθούν με αυτού του είδους τις νομικές πράξεις να περάσουν και από τη δική μας και με τη δική μας συμμετοχή. Μπορεί να σκεφτεί λοιπόν η Επιτροπή τι θέλει. Θέλει ευελιξία με τη μορφή η οποία ουσιαστικά θα μας συμπεριλαμβάνει και στο πρόγραμμα εργασιών και στις κατεξουδιοδότηση πράξεις, είτε θέλει ουσιαστικά και στην υλοποίηση να μας συμπεριλαμβάνει. Εμείς σε κάθε περίπτωση σαν νομοθετική αρχή πρέπει να θέτουμε τις προτεραιότητες και η Επιτροπή πρέπει να επιλέξει τι ακριβώς θέλει. Η Επιτροπή γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο με τις πράξεις αυτές όταν ουσιαστικά συμπεριλαμβάνουν καθαρά θέματα υλοποίησης προγραμμάτων, τεχνικής υλοποίησης των προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ, Σίλβια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και ευχαριστώ και την Πέτρα διότι ε, η Κριστίν Λιμπάτσκι έκανε ε, εξαιρετική εργασία, αλλά δυστυχώς ε, δεν, μπορεί να βρίσκεται μεταξύ μας και αυτό προσφέρθηκα να την αντικαταστήσω. Θα ήθελα να πω ότι πίστευα ότι δεν έχει κλείσει η συζήτηση. Το θέμα αυτό είναι ύψης της σημασίας για όλες τις ομάδες. Θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα οι σε προοπτικές τριπλασιασμού των ε, ταμείων και των κονδυλίων αφορά μια καλύτερη ενσωμάτωση και Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι το, θέμα των λιγότερων ευκαιριών αφορά και εκείνους που προέρχονται από ένα μεταναστευτικό περιβάλλον, ε, αμαία και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν λιγότερες ευκαιρίες ε, συμμετοχής στα προγράμματα κινητικότητα. Το Erasmus Mundus έχει επανεισαχθεί και χαίρομαι γιατί το δέχτηκαν πολύ όχι μόνο οι σοσιαλιστές. Εδώ μιλάμε και για διδακτορικά αλλά και για μάστερ. Στο, ως προς το Discover You θεωρούμε ότι το θέμα αυτό, το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα και έχουν υποβληθεί τροπολογίες έτσι ώστε να υπάρχει μία εκπαιδευτική περισσότερο διάσταση. Και επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει εγκάρσιος χαρακτήρας ε, μαζί με άλλα προγράμματα θα δούμε πώς θα οριστούν οι συμβιβαστικές. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα digital αλλά και που άπτονται του πολιτισμού. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μία συνεργασία μέσα στα πλαίσια των εταιρικών ε, σχέσεων γιατί εδώ μιλάμε για εταιρικές σχέσεις όχι μόνο μέσα στα πανεπιστήμια. Ως προς τις προοπτικές μεγαλύτερες ευελιξίας μετά τα διπλώματα, για να μπορεί κανείς ε, να έχει ένα-δύο χρόνια περισσότερο, αυτό το είδαμε στα μεγάλα οδεία και ούτω καθεξής θα πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης έχουμε κινητοποιηθεί σε πολλά μέτωπα. Θα πρέπει να επανεισάγουμε προγράμματα ψηφιακών διαρθρώσεων και δομών τύπου blended και θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα ε, εξελιχθούν οι σχέσεις Συμβουλίου-Κοινοβουλίου. Όταν αλλάζουν οι πολιτικές ε, προτεραιότητες, είναι σαφές ότι θα πρέπει να εμπλέκεται και το Κοινοβούλιο. Ο Λουίτσι Μόργανο. Ευχαριστώ. Εντάχει. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν είχα τις τροπολογίες, δεν τις είδα. Γι' αυτό δεν μπορώ να ε, μιλήσω επί της ουσίας. Ε, μιλώ για τις συμβαστικές. Δυστυχώς ε, διανεμήθηκαν την Παρασκευή και δεν τις έλαβα. Θα ήθελα να παρέμβω ως προς το εξής. Ως προς την επαγγελματική κατάρτιση ο εισηγητής μας επισύρει την προσοχή σε αυτές τις δυνατότητες, επιπλέον δυνατότητες του Εράσμους και μιλά για εμβάθυνση του ζητήματος όπως έχει γίνει από την Επιτροπή μας. Για να λάβουμε υπόψη την κωδικοποίηση που υπάρχει στις διάφορες χώρες. Επίσης, θα ήθελα να μου πει ο εισηγητής πώς σκέφτεται ως προς τον ε, κανονισμό Εράσμους γίνεται λόγος για διαπολιτισμικό διάλογο σε σχέση με την νεότητα. Και, αλλά δεν γίνεται λόγος για θρησκευτικό διάλογο, διάλογο δηλαδή μεταξύ των διαφόρων ε, θρησκευμάτων. 15-18. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούμε αυτό το θέμα για τους ίδιους λόγους που προανέφερα θα ήθελα να δοθεί μια απάντηση σε αυτό έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ως προς τις αρχές της ανεξιθρησκείας. Και υπάρχει και το θέμα της συνθήκης, το άρθρο 22 τη, του χάρτη των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων και γι' αυτό αναφέρομαι σε βασικά κείμενα, τα οποία δεν από τα οποία δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε. Ωραία. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ο Μίλαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με αυτό που μόλις είπε ο κύριος Μόργαν, Η τροπολογία σας από ό,τι μου λένε είναι μέσα στο κείμενο για το θρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο έχουν συμπεριληφθεί. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα, λογικά. αλλά από ό,τι βλέπω, εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά αρκετά ζητήματα. Έχουμε καταλήξει συμφωνία πράγματι για αρκετά. Και θα διαπραγματευτούμε και με τις άλλες ομάδες, αλλά έχουμε ακόμα κάποια ζητήματα ανοιχτά. Γι' αυτό και έχουμε δύο ε, ήδη συναντήσεις ε, σκιωδών και τρεις συναντήσεις με τους εμπειρογνώμονες και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτά τα διλήμματα. Γιατί υπάρχουν σίγουρα κάποια επίμαχα θέματα, αλλά πιστεύω πως θα καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Δεν θα είναι κανείς μας ισχυρογνώμων. Όλοι θα δείξουν επικοδομητική στάση στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου αλλά σε ό,τι αφορά κάποια βασικά ζητήματα, σίγουρα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία, να καθίσουμε γύρω από το δύο τραπέζι και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Και οι εμπειρογνώμονε ελπίζω και αυτοί να μπορέσουν μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους. Να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις ή σχόλια αλλά δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν και σκόπιμο να το κάνω σήμερα, γιατί έχουμε και αύριο συνάντηση των εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Προστατεμένη Αξία είναι μια τυπική προσέγγιση για όλα τα προγράμματα και για όλες τις νομοθετικές πράξεις. Είναι μια καλή έννοια. Μας βοηθά να αξιολογήσουμε τα προγράμματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την εκπαίδευση, την νεολαία, το εράσμους, ήπια προσέγγιση κυρίως. Δηλαδή δύσκολα μπορεί κανείς να βρει ε, μια ποσοτικοποιημένη αξιολόγηση για να τα συμπεριλάβουμε σε, κάποιο, σε διάγραμμα τα στοιχεία για παράδειγμα. ενιολογικά πρέπει να το δούμε. Η ευρωπαϊκή προστάμενη αξία βέβαια κάπως πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θέλουμε το Εράσμους να το διαχωρίσουμε από το τοπικό ή το εθνικό επίπεδο, όχι. Απλά μιλάμε για μια προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση. Δεν έχει να κάνει με τεχνικής φύσεω προσέγγιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ίδια ε, ίση αμοιβή για ίδια εργασία, φυσικά ε, πρέπει να το τονίσουμε, δεν διαφωνώ. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά βέβαια πρέπει να μιλήσουμε και για τον προϋπολισμό. Και αυτό θα είναι ένα πιο δύσκολο θέμα, γιατί έχουμε και τα άλλα θεσμικά όργανα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Συχνά ακούμε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση, στην νεολαία, είναι καλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ευρέως διαδεδομένη έννοια και ελπίζω και ε, στις διαβουλεύσεις να το καταλάβουν και οι συνομιλητές μας. Σας ευχαριστώ για τα σχολιά σας. Ε, τώρα βλέπω και που έγκυνται οι διαφωνείς. Ανησυχώ κάπως βέβαια, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Ευχαριστώ. Μήπως σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι βεβαία ότι θα τα καταφέρουμε με πνεύμα ομαδικότητας και κοινού νου. Θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε συμβιβαστικέ προτάσεις. Και εγώ περιμένω να δω πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες. Εγώ νομίζω ότι πιο δύσκολη θα είναι η διαβούλευση με το Συμβούλιο παρά εμείς εδώ το πώς θα τα βρούμε μεταξύ μας. Εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι το δυνατόν για να βρούμε ως το τον καλύτερες συμβαστικές προτάσεις που θα ε, βρουν σύμφωνοι στο τέλος να στο δυνατόν μεγαλύτερη πλειονότητα των συναδέλφων. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης ήδη στα διάφορα δεν βλέπω αν θέλει κάποιος το λόγο Άρα το μόνο που μου απομένει να κάνω να σας πω ότι 21 Ιανουαρίου, τις 3 μέχρι τις 6.30 ημέρα Δευτέρα και 22 Ιανουαρίου όλη τη μέρα την Τρίτη, 1 με 12.30 και 3 με 6.30, είναι η επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστεί η Πρόεδρος τους Διερμηνής και καλά Χριστούγεννα σε όλες και όλους. Και τους περισσότερους θα σας δω και την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Γεια σας.